Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να καθυστερούν λόγω περίοδου πρώτων καλοκαιρινών διακοπών, αλλά ας ξεκινήσουμε με την έγκριση της σημερινής διάταξη. Έχω μία αλλαγή να σας ανακοινώσω. Σήμερα το πρωί, στο τέλος της συνεδρίασης, μετά την ε, ε, συζήτηση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την Ελλάδα, έχουμε ένα πρόσθετο σημείο προετοιμασία της συνεργασίας με την Ερυθρέα. Το σημείο αυτό θα γίνει και των θυρών μετά το τέλος της κοινή συνεδρίασης με τη ΛΥΜΠΕ. Οπότε μετά τις, ε, τη συνάντηση αυτή, όποιος ε, πρέπει να φύγει, παρακαλώ να αποχωρήσει από την αίθουσα. Ίσως να συνεχίσει μέχρι τη μία αυτό το σημείο, αλλά χωρίς διερμηνία μετά τις 12.30. Εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε με τα άλλα σημεία της μερίσιας διάταξης. Μπορούμε να εγκρίνουμε την μερίσια διάταξη με αυτή τη μία τροποποίηση. Ωραία, εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Έχω μία μόνο ανακοίνωση ότι δεν έχουμε διερμηνία στα σλοβακικά σήμερα το πρωί Ζητούμε συγγνώμη για όσου θα ήθελαν διερμηνία στα σλοβακικά. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών προηγουμένων συνεδριάσεων. Συνεδρίες της Επιτροπής 29 και 30 Μαΐου. Αν έχετε παρατηρήσεις, παρακαλώ να τις κοινοποιήσετε στη γραμματεία πριν το τέλος της συνεδρίασης. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θα θεωρούνται ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Σημείο 4. Ανακοινώσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πει κάτι? Όχι. Οπότε Περνάμε στο σημείο 5. Εδώ έχουμε προκαταρκτικά ευρήματα της ε, αξιολόγησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε συναδέλφους από την Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, και η Πρόεδρος κυρία Βαλεάν είναι μαζί μας σήμερα το πρωί, διότι ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας αφορά και τις δύο επιτροπές και τα 28 κράτη-μέλη, συν την Ισλανδία, Νορβηγία, Σερβία, Φυρό, Μοντενέγρο και Τουρκία, συμμετέχουν στο Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται για ένα μηχανισμό ε, προειδοποίηση σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, ε, πλημμύρας ε, ή κρίσεων όπως η κρίση του έμπολα στη Δυτική Αφρική ναι. Συγκρούσει στην Ανατολική Ουκρανία και στο Ιράκ, ε, κρίση ε, όπως το προσφυγικό και άλλα. Ε, υπάρχει το Κέντρο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, Κέντρο Συντονισμού της Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών, το οποίο ε, λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, ε, ε, ακόμη και στις γιορτές των Χριστουγέννων, λίγο πιο, λίγους δρόμους πιο μακριά από εδώ, στην Λελουά, και πρόσφατα επισκεφτήκαμε τις εγκαταστάσεις τους όταν μας κάλεσε ο Επίτροπος Τηλιανίδης. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας υπόκειται στον κανονισμό τον οποίο γίναμε το 2013 αξιολογείται και σήμερα το πρωί θα ακούσουμε κάποια από τα ευρήματα αυτής της ε, αξιολόγησης. Θα δώσω όμως το λόγο στην κυρία Βαλέαν πριν να συνεχίσω. Ευχαριστούμε κυρία Μακάβαν. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε σε αυτήν την κοινή ανταλλαγή απόψεων. Εκ μέρους της Επιτροπής ΕΝΒΗ χαιρετίζω αυτή τη σημερινή συνεδρίαση και την ευκαιρία που μας δίνεται. Όπως είπατε, η αντιπροσωπεία της Επιτροπής ΕΝΒΗ επισκέφθηκε το Κέντρο Συντονισμού της Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών κατόπιν προσκλήσεως του Επιτρόπου Στυλιανίδη στις 30 Μαΐου. Το κέντρο αυτό είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα της προστιθέμενης αξίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μας βοηθάει να αποφεύγουμε περί επικάλυψη ε, προσπαθειών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών σε ολόκληρο τον κόσμο. Κατά την επίσκεψή μας αναφέρθηκαν ορισμένες ανησυχίε για το διαθέσιμο προπολογισμό και για την ανάγκη να βρεθούν λύσεις για καταστάσεις οι οποίες επιβαρύνουν ιδιαίτερα κάποια κράτη-μέλη. Παραδείγματο χάρη, καταστάσεις τις οποίε απαιτούνται απαιτείται βοήθεια ε, ιατρικού περιεχομένου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ε, η ενδιάμεση αξιολόγηση θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο από την Επιτροπή για ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία της υλοποίηση των προηγουμένων αποφάσεων και πρέπει να ε, υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου. Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί η ενδιάμεση έκθεση αξιολόγησης. Ελπίζουμε όμως σήμερα ότι θα ακούσουμε κάποια σημαντικά στοιχεία, ιδίως το αποτέλεσμα της ανοιχτής διαβούλευσης που οργανώθηκε από την Επιτροπή. Αν μου επιτρέπετε, θα δώσω απευθείας το λόγο στον Διευθυντή εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Ιωάννη Λούχνε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Βαλεάν, αγαπητοί συνάδελφοι. Ξεκινώ ζητώντα συγγνώμη για την ημερομηνία που αναφέρατε, γιατί είπατε ότι μέχρι τέλος Ιουνίου έπρεπε να έχει υποβληθεί η έκθεση και έχει περάσει αυτή η ημερομηνία. Αυτό έχει σχέση με τη διαδικασία αξιολόγησης, διότι τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία πήραμε αφορούσαν την ποιότητα και δεν ήταν πολύ ικανοποιητικά τα ευρήματα. Ζητήσαμε λοιπόν από τους αξιολογητές να διαβρύνουν την έρευνά τους. Γι' αυτό καθυστερήσαμε και γι' αυτό δεν έχουμε ακόμη την τελική αξιολόγηση. Πολύ σύντομα θα την έχουμε όμως. Και το Σεπτέμβριο θα ε, έχετε την έκθεση αντί το, του Ιουνίου που αρχικά έπρεπε να είναι έτοιμη θα ήθελα να παρουσιάσω την τρέχουσα κατάσταση στους τρεις τομείς ε, δραστηριότητα, ε, ετοιμότητα, πρόληψη και ε, ανταπόκριση και να πω και ποιες είναι οι προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε. Αυτά τα οποία θα σας πω δεν διαφωνούν με αυτά τα οποία έχω δει ως προκατακτικά ευρήματα της έκθεσης, αλλά έχουμε και μια έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου και υλοποιούμε τα συμπεράσματά τους και υπάρχει και μια συνεχής διαδικασία ανατροφοδότησης, οπότε τα διδάγματα τα οποία αποκομίζουμε προσπαθούμε να τα εφαρμόζουμε στην πράξη. Γενικά, υπάρχει συνένεση ότι η απόφαση για ένα μηχανισμό πολιτικής προστασίας, αυτή που ελήφθη το 2013, λειτουργεί σωστά. Τώρα είμαστε στον τέταρτο χρόνο υλοποίησης και τα συνολικά αποτελέσματα θεωρώ ότι είναι ικανοποιητικά διότι ο μηχανισμός θεωρείται βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος που είχαμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ετοιμότητα, πρόληψη και ανταπόκριση φυσικών καταστροφών. Για την πρόληψη, η καινοτομία είναι ότι σύμφωνα με την νομοθεσία πρέπει να γίνεται εθνική αξιολόγηση και από τα 28 κράτη-μέλη, αξιολόγηση κινδύνων, ε, λάβαμε την αξιολόγηση αυτή και παρατηρούμε ότι σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν άλλα υπουργεία και άλλοι οργανισμοί εκτός ε, του Υπουργείου που είναι αρμόδιο για την πολιτική προστασία και με βάση τις εκθέσεις των κρατών μελών ε, διαμορφώσαμε μια συνολική έκθεση κινδύνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση που παρουσιάζει το συνολικό πεδίο των κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά υποστηρίζονται με ένα σημαντικό προϋπολογισμό για την πρόληψη και πρέπει να τονίσω ότι για την ετοιμότητα και την πρόληψη δαπανούμε πολύ μεγαλύτερο ποσό από ότι για την αντιμετώπιση των κινδύνων για την ετοιμότητα και αυτό νομίζω ότι είναι και η κύρια καινοτομία του κανονισμού έχουμε την ικανότητα άμεσης αντιμετώπισης αυτό εμείς το αποκαλούμε ε, εκούσια ε, συγκέντρωση πόρων δηλαδή τα κράτη-μέλη εκουσίως συνεισφέρουν πόρους ε, σε μια κοινή δεξαμενή πόρων και για τα περισσότερα τμήματα με τα οποία ασχοληθήκαμε, οι πόροι μας ε, ε, υπερέβησαν ε, τους αρχικά διαθέσιμους πόρους. Και συνολικά έχει βελτιωθεί η ποιότητα των πόρων μας. Έχουμε και δύο συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία μπορείτε και να δείτε στο κέντρο. Υπάρχει το Ευρωπαϊκό Σύστημα προειδοποιήσεις για τις ε, ε, πλημμύρες. Αυτό βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα ε, όσον αφορά τις βροχοπτώσεις και είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο προβλέψεων για το πού μπορεί να συμβεί κάποια πλημμύρα. Και έχουμε και το σύστημα πληροφόρησης για τις πυρκαγιές, δυστυχώς πολύ επίκαιρο αυτές τις μέρες, και είναι εργαλεία τα οποία διατίθεται και για τα 34 κράτη που συμμετέχουν. Έχουμε επίσης μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, η υπηρεσία χαρτογράφησης μετά μια καταστροφή που βασίζεται στο σύστημα Κοπέρνικους, διότι δεν δίνουμε μόνο χάρτες, αλλά δίνουμε χάρτες που έχουν και ένα επιπλέον στοιχείο μετά τις αναλύσεις που έχουν γίνει, ώστε αυτό δίνει περισσότερα στοιχεία σε αυτούς που παρέχουν ε, βοήθεια κατά τη διάρκεια κρίσεων, ε, καθώς και αναλυτικά δεδομένα μετά την παρέμβαση. Κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό στη δημιουργία ε, ευρωπαϊκής ικανότητας ενός ευρωπαϊκού σώματος είναι η εκπαίδευση. Τα τελευταία τρία χρόνια διπλασιάσαμε τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων. Έχουμε 740 το χρόνο, ενώ προηγουμένως είχαμε 322 εμπειρογνώμονες το χρόνο. Το 50% μόνο είναι γυναίκες και αυτό οφείλεται και στο επάγγελμα αλλά και στη χώρα προέλευσης των ατόμων. Ε, είναι ένα ποσοστό το οποίο θα θέλαμε να διατηρείται υψηλό. Για την ε, ετοιμότητα το διαθέσιμο κονδύλι είναι 17 εκατομμύρια ευρώ. Το 2014 και 2015 ο μηχανισμός ενεργοποιήθηκε 19 φορές το χρόνο. Το 2016 ενεργοποιήθηκε 26 φορές. Η τάση λοιπόν είναι ανωδική. Και για να σας δώσω μια εικόνα, από το 2014 μέχρι το 2016, περίπου 33% των ετοιμάτων προήλθαν από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα υπόλοιπα 2 τρίτα από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο και τα Ηνωμένα Έθνη μπορούν να ζητήσουν βοήθεια στην οποία εμείς κρίνουμε αν θα ανταποκριθούμε, αλλά ούτω ή άλλω ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη για τα αιτήματα που λαμβάνουμε. Είναι ενδιαφέρον λοιπόν ότι η δραστηριότητά μας είναι εντονότερη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παρά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα περνώ στην έρευνα που κάναμε και στα ερωτήματα που θέσαμε. Τα τρία τέταρτα των αρχών πολιτικής προστασίας θεώρησαν τις διαδικασίες συντονισμού έγκαιρες ε, και ε, ομαλές. Όσον αφορά τις προκλήσεις, ε, το βασικό θέμα που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αλλάζει το φάσμα των κινδύνων. Τώρα περισσότερο έχουμε κατά νου την ανταπόκριση σε προβλήματα τρομοκρατίας αντιμετώπιση ε, βιολογικών, πυρηνικών ε, και λοιπόν κινδύνων ε, έχει λάβει μεγαλύτερη προτεραιότητα. Οι κυβερνοεπιθέσεις επίσης μας αφορούν, διότι αν υπάρξει μία επίθεση στο σύστημα επικοινωνιών του κέντρου συντονισμού δεν θα λειτουργεί σωστά σε περίπτωση δηλαδή, που υπάρχει μια επίθεση που εξουδετερώνει τη σύνδεσή μας στο διαδίκτυο. Όσον αφορά την πρόληψη και την ετοιμότητα, φιλοδοξούμε να εστιάσουμε περισσότερο τις δράσεις μας στο μέλλον. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για ετοιμότητα και πρόληψη προέρχεται από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείο Συνοχής και ο προϋπολογισμός μας ε, είναι πολύ μικρός. Ε, θέλουμε λοιπόν να εντείνουμε τις συζητήσεις με τις εν λόγω γενικές διευθύνσεις και με τα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε πώς ακριβώς χρησιμοποιούνται τα κονδύλια και αν ε, αυτά τα οποία γίνονται βασίζονται στην ανάλυση κινδύνων. Για την ετοιμότητα Ε, υπάρχει μια ιδιαίτερα ποιοτική διαδικασία, η οποία όμως είναι αρκετά χρονοβόρος για την καταγραφή των διαδικασιών και θέλουμε ε, να, να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τη διαδικασία. Αυτό το οποίο ε, επανέρχεται στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη και όλους τους άλλους είναι ότι η απόφαση δημιούργησε μηχανισμούς οι οποίοι σε ορισμένους τομείς είναι κάπως γραφειοκρατικοί με το παρόν πλαίσιο ήδη μπορούμε να κάνουμε πολλές δράσεις και προσπαθούμε να βελτιώσουμε τη δράση μας. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα όσον αφορά την αντιμετώπιση αναγκών. Έχουμε ένα σύστημα συγχρηματοδότησης των μεταφορών όπου προς το παρόν λαμβάνουμε εγγράφος τις αιτήσει και εγγράφος τα τιμολόγια και μερικές φορές τα τιμολόγια τα παίρνουμε τόσο αργά που είναι δύσκολο να κάνουμε τη διαχείριση του προϋπολογισμού μας. Βάσει των συστάσεων του ελεγκτικού συνεδρίου, μέχρι το τέλος του επομένου έτους θα φροντίσουμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο θα βασίζεται στην πληροφορική, θα είναι ένα μηχανογραφημένο σύστημα και δεν θα βασίζεται σε χειρόγραφα στοιχεία και ε, θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα του αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανονισμού και να απλουστεύσουμε το σύστημα πληρωμών, ούτω ώστε όταν στείλουμε ένα αεροπλάνο από τη Γαλλία στην Πορτογαλία να ξέρουμε ήδη πόσο κοστίζει και να έχουν συμφωνήσει και οι δύο πλευρές. Προσπαθούμε λοιπόν να μειώσουμε τη γραφειοκρατία. Όσον αφορά την ανταπόκριση, Κατά τις συζητήσεις με το ελεγκτικό συνέδριο έχουμε πει ότι θα καταγράφουμε και έχουμε ένα σύστημα καταγραφής αυτή τη στιγμή για όλες τις δράσεις του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας για να μπορέσουμε να μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα για τις πυρκαγιές στη Χιλή, παραδείγματο χάρη, χρειαστήκαμε 48 ώρες ακριβώς από τη στιγμή που λάβαμε το αίτημα μέχρι ότου επιτόπου βρέθηκαν 200 ε, πυροσβέστες ε, στη Χιλή για την αντιμετώπιση των ε, πυρκαγιών. Ο χρόνος απόκρισης ήταν από μισή μέχρι μια μισή ώρα από τη στιγμή που λαμβάνουμε την αίτηση μέχρι που στέλνουμε τη βοήθειά μας. Είναι λοιπόν αποτελεσματικός ο χρόνος ε, ανταπόκρισής μας. Τώρα, για το τι γίνεται από εδώ και πέρα. Κάνουμε συζητήσεις με όλους τους εμπλεκομένους φορείς και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε στο πλαίσιο το τωρινό, δηλαδή προσπαθούμε να μην ε, καθυστερούμε, να μην μένουμε άπραγοι, αλλά να βελτιώνουμε την αποτελεσματικότητά μας συνεχώς. Δεν θα προτείνουμε κάποιες αλλαγές στην απόφαση τώρα, αλλά θα κάνουμε μία εις βάθος συζήτηση με τα κράτη-μέλη, κάτι που το κάνουμε ήδη, αλλά εδώ θα γίνει πιο συγκεκριμένα για να ε, λάβουμε υπόψη τα κράτη-μέλη και αυτά τα οποία έχουν να μας πούν για την υποστήριξη που χρειάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την επισκόπηση της ε, κατάστασης. Νομίζω ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού συζητά σχετικά θέματα σήμερα ή θα τα συζητήσει στο τέλος της πρωινής συνεδρίασης. Ο κύριος Νόιζερ πρώτα. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίαση. Συνολικά νομίζω ότι η παρουσίασή σας δείχνει ε, θετικές εξελίξεις. Έχω μία ερώτηση για την κλιματική αλλαγή. Είπατε ότι εν των μέσων, εν των πόρων ε, χρησιμοποιούνται στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν σχέση με την αλλαγή του κλίματος αυτοί οι πόροι που διατίθενται. Μια δεύτερη ερώτηση για την κυβερνοασφάλεια. Υπήρξαν ε, περιστατικά στα οποία δέχθηκατε κάποιες απειλές για το κέντρο συντονισμού, ε, υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες συνεισφέρατε για κύβερνο επιθέσεις. Και μια τρίτη ερώτηση για τη διαχείριση κινδύνων. Στην έκθεσή σας ε, καταγράφονται ορισμένε χώρες όπω το Νεπάλ ή χώρες της Δυτικής Αφρικής που επλήγησαν από τον ε, έμπολα. Σε τέτοιες χώρες πόσο ε, παραμένουμε ε, και παρέχουμε βοήθεια στο πλαίσιο της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ε, και πότε αρχίζουν να παρεμβαίνουν οι υπηρεσίες που αρμόδιες για την ανάπτυξη. Πώς γίνεται δηλαδή η διαχείριση κινδύνων. Και τελευταία ερώτηση. Η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ασχολείται με ε, τα δικά σας μέτρα αντιμετώπισης ή είναι περισσότερο επαγγελματίες οι οποίοι ασχολούνται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και εγώ είχα κάποιες ερωτήσεις για την κυβερνοασφάλεια, η οποία είναι ένα ζήτημα που αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία. Ε, σκέφτεστε να υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα. Και όταν ανέλαβα ε, την Προεδρία αυτής της Επιτροπής πριν ε, το ξέσπασμα της κρίσης του έμπολα, είχαμε συζητήσει ε, για την ε, μεταφορά των υπηκών Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα μεταφέρονταν ενώ είχαν ε, προσβληθεί από τον ιό έμπολα και ποιος θα χρηματοδοτήσει αυτή την μεταφορά. Υπήρχαν και σκέψεις, ήταν κάτι το εξαιρετικά ακριβό. Έχει λυθεί αυτό το ζήτημα της εκένωσης, αν θέλετε, του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τέτοια μέρη σε επίγουσα περίπτωση. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ. Λέει ο κύριος Λούχνερ, για να απαντήσω στο αξιότιμο μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Νόιζερ, να σας πω ότι όταν μίλησα για το 1 τρίτο των μέτρων, εννοούσα το 1 τρίτο των απαντήσεων. Ε, από επιστημονική σκοπιά δεν μπορώ να τα συσχετίσω άμεσα με την κλιματική αλλαγή. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι εξ όσων θυμάμαι, η μεγάλη πλειοψηφία πάνω από το 90% με εξαίρεση την μετανάστευση είναι περιστατικά που σχετίζονται με εθνικές καταστροφές, με πλημμύρες, με πυρκαγιές, δασικές. Ε, από τη στατιστική γνωρίζουμε ότι και στην περίπτωση των πυρκαγιών και στην περίπτωση των ε, πλημμύρων τα τέτοια γεγονότα είναι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο ακραία τα φαινόμενα και οι, οι θερμοκρασίες αυξάνονται. Επομένως, προσωπικά Απαντώ ναι. Προσωπικά πιστεύω ότι η κλιματική αλλαγή είναι κάτι που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, όχι μόνο ως προς τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε στη κρίση, αλλά κυρίως ως προς τη δυνατότητα να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι και να κάνουμε πρόληψη, να προλάβουμε. Είναι δύσκολο βέβαια να γίνουν όλα αυτά, γιατί υπάρχουν και πολιτιστικές παραδόσεις, συμφέροντα της κοινωνίας, οικονομικά συμφέροντα, κράτη που πρέπει να προσαρμοστούν και να προσαρμογή ορισμένη αλλαγή και κάποιες από τις αλλαγές που απαιτούνται είναι πραγματικά πολύ βαθιές, αλλά θεωρώ ότι τέτοιου τους φαινόμενα στην πλειονότητά τους συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Τώρα, γιατί η κυβερνοασφάλεια και το κατά πόσο είμαστε προετοιμασμένοι. Έχω να πω τα εξή. Γνωρίζετε ότι είναι δυνατό να σταματήσει ο πυρηνικός ε, εμπλουτισμός επιτόπου με έναν ιό. Ε, θεωρητικά είναι αυτό εφικτό. Εάν μπορεί κανείς να αλλάξει τα ε, ε, GSM, τα σήματα, τότε μπορεί να αποκόψει το ρεύμα από μια ολόκληρα η πόλη και να τη βυθίσει στο σκοτάδι. Νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι και προετοιμαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διάφορες χώρες δαπανούν σημαντικά ποσά, έχουν αυξημένους προϋπολογισμούς και έχουν να κάνουν με χιλιάδες ανθρώπους που ενισχύουν την κυβερνοασφάλεια κυρίως στο στρατιωτικό και αμυντικό τομέα. Εμείς έχουμε ένα περιστατικό και έτσι απαντώ και στην ερώτηση της Προέδρου. Ε, ε, είχαμε ένα περιστατικό όπου δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι ακριβώς ήταν, αν ήταν επίθεση ή όχι, αλλά σταμάτησε το διαδίκτυο να λειτουργεί και το σύστημα το πληροφοριακό μας βασίζεται στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο. Δεν νομίζω ότι το σύστημα μπορεί να δεχθεί εύκολη επίθεση από μόνο του γιατί είναι αυτόνομο αυτούσιο και ασφαλές, δεν είναι ανοιχτό για, ε, σε δράσεις επιτόπου, field operations. Και είναι μια συζήτηση που κάνουμε με τα κράτη-μέλη, πώς διασφαλίζουμε ότι όσοι ενεργούν επί τόπου έχουν ε, ακριβείς πληροφορίες, αφού το σύστημα είναι μόνο ανοιχτό σε εμά και όχι σε όσους δραστηριοποιούνται επί τόπου αλλά εν πάση περιπτώσει είναι αυτός ένας τομέας στον οποίο πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, αλλά και ο ιδιωτικό τομέας πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα και αυτό πρέπει να το πούμε. Είναι ένας τομέας πολύ ενδιαφέρον γιατί έχουμε και υβριδικές απειλές. Αυτό το θέμα μας έρχεται από το ΝΑΤΟ, γιατί το ΝΑΤΟ ανησυχεί όλο και περισσότερο για όλα αυτά. Ως προς τη διαχείριση κινδύνου τώρα θα έλεγα για την και όχι το ΝΑΤΟ, σε πάση περιπτώσει στη διαχείριση κινδύνου ε, λόγω της γεωγραφικής θέσης της ΑΕΤΗΣ και, της, ε, ε, και των καταστάσεων εκεί. Έχουμε συμβάντα κάθε δύο χρόνια, είναι συνεχής ο διάλογος. Όταν συναντήσαμε την αντιπροσωπεία της ΑΕΤΗΣ στην Κανκούν, είπαμε ξεκάθαρα ότι με χαρά να αποστείλουμε συμβουλευτική αποστολή, αλλά εν πάση περιπτώσει πρέπει και αυτοί να ψηφίσουν ένα νόμο πολιτικής προστασίας. Ε, είναι μια υπόσχεση που μας έχουν δώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν την έχουν εκπληρώσει, τελικά πρέπει να το κάνουν, γιατί βασικά αυτό που χρειάζεται στη χώρα είναι η αποκέντρωση ορισμένων αρκετών εξουσιών και η ύπαρξη τοπικών θεσμών πολιτικής προστασίας έτσι ώστε όταν συμβεί μια καταστροφή να υπάρχει δυνατότητα μια τοπική ομάδα να ανταποκριθεί άμεσα. Αυτός ο νόμος δεν έχει ψηφιστεί ούτε καν πριν από μια-δύο εβδομάδες ακόμα που το κοίταξα τελευταία φορά. Επομένως, εμείς δίνουμε συμβουλές, κάνουμε ανάλυση και την οποία αναλαμβάνει και υιοθετεί η αναπτυξιακή συνεργασία. Η, DG, η Γενική Διεύθυνση ΤΕΦΚΟ είναι πολύ ενεργή, για παράδειγμα, με τις χώρες ΑΣΕΑΝ, αλλά χρειαζόμαστε πιο σοβαρούς συνεταίρους και ομολόγους στην ΑΕΤΗ. Τώρα, ε, η απάντηση είναι όχι ακόμα για το κατά πόσο θα υπάρξει εθελούσιο και εθελοντικό σώμα. Υπάρχει πρόταση για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό οι αρχές για την πολιτική προστασία και είχαμε σκεφτεί να δραστηριοποιούνται στους τομείς της προετοιμασίας, της ετοιμότητας και της πρόληψης. Κάθε χρόνο, τον Απρίλιο και τον Μάιο, είναι πάρα πολλές οι εκτάσεις που είναι καλό να καθαριστούν τα, χλαμό, τα χαμόκλαδα, ακριβώς για να είναι καθαρό το έδαφος και να μειωθεί η πιθανότητα πυρκαγιά στη συνέχεια το καλοκαίρι. Είναι τεράστια, τεράστιες οι εκτάσεις αυτές, χρειάζεται η βοήθεια των εθελοντών και θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση στο σώμα αλληλεγγύης και στο σώμα εθελοντών που θα βοηθούσαν για αυτές τις δραστηριότητες. Τώρα για το Μεντεουάκ, Έχουμε τέτοιου είδου δυνατότητες στο σώμα των εθελοντών, αλλά για τις ε, ε, υψηλά μεταδοτικές και λοιμώδεις ε, νόσους όπως ο έμπολα η απάντηση είναι όχι. Να σας δώσω το παράδειγμα του Λουξεμβούργου, το οποίο μας έδωσε ένα αεροπλάνο, πλήρωσε αυτό το αεροπλάνο για τη διαχείριση της κρίσης του έμπολα και μας είπε το Λουξεμβούργο που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να χρηματοδοτούμε τη συντήρηση αυτού του εργαλείου χωρίς να το χρησιμοποιούμε και χωρίς εισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι λογικό. Ένα από τα σημεία που συζητείται μεταξύ των κρατών μελών πάντοτε είναι και αυτό το ερώτημα που θέσατε εσείς στην αρχή. Ε, πώς γίνεται η συγχρηματοδότηση και με ποιο σκοπό, με ποιους σκοπούς. Επομένως, εμείς δεν χρηματοδοτούμε τα αεροσκάφη MetaWAC. Και άρα πάρα πολλά ε, στοιχεία ενεργητικού που θα μπορούσαμε να έχουμε παραμένουν εκτός συστήματος. Επομένως έχουμε μία βασική δυνατότητα ε, ε, κένωσης για τις ε, ψηλά λοιμώδεις ασθένειες. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ. Πράγματι, είναι πρόβλημα αυτό. Ήταν και την προηγούμενη φορά. Φαινόταν ότι είναι σχετικά εύκολο να λυθεί αυτό το ζήτημα. Δυστυχώ το Συμβούλιο δεν μπόρεσε να το λύσει. Παρακαλώ. Κάνεν Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας και ευχαριστούμε για την ε, εισαγωγική σας παρουσίαση. Μας δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφθούμε επιτόπου τις εγκαταστάσεις ε, του ERCC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Συντονισμού Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών και είδαμε ότι όλα λειτουργούν ε, πάρα πολύ καλά. Μία ερώτηση θα ήθελα να κάνω. Μία από τις συστάσεις του ελεκτικού συνεδρίου ήταν να εξετάσετε μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αντιμετώπισης ε, Λοιμόξεων ε, τι διατάξεις θα απαιτούνταν, ούτως ώστε να χρησιμοποιούνται και οι εμπειρογνώμονες του ECDC σε περίπτωση καταστροφών. Έχουν γίνει κάποια βήματα, πώς βλέπετε την κατεύθυνση των ε, πραγμάτων. Χρειάζεται υποστήριξη από το, από το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ναι, για την ερώτηση αυτή θέλω να πω ότι το συζητάμε στις, ε, με τις διάφορες γενικές διευθύνσεις, γιατί το πρόβλημα είναι η εντολή που έχει ο οργανισμός. Θα πρέπει να γίνει κάποια τροποποίηση. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου του ECDC, αλλά κρίνοντας από τη συμμετοχή τους στις δικές μας δράσεις, νομίζω ότι ενδιαφέρονται. Χτες και προχτές κάναμε μία διήμερη συνεδρίαση με το Αμερικανικό Κέντρο ε, Ελέγχου νοσημάτων και συμμετείχαν και το ECDC και η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με την αποστολή εμπειρογνωμόνων, γιατί έχουν 20.000 εμπειρογνώμονες, δηλαδή ένα δυναμικό που θα μπορούσαμε και που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Γενικά όλοι συμφωνούμε ότι θα ήταν καλό να συμμετέχει με πιο εύκολο τρόπο το ECDC αλλά ε, απαιτείται τροποποίηση της εντολής και αυτό σημαίνει και αντίστοιχους πόρους. Δηλαδή η συζήτηση βρίσκεται εν εξελίξη αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι συγκεκριμένα σχεδιάζει η Γενική Διεύθυνση για θέματα υγείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Φρουντζουλίτσα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον προσκεκλημένο μας η συνεργασία πώς γίνεται με χώρες που δεν είναι μέλη με της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Μαυροβούνιο, η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, η Τουρκία, η Σερβία. Ποιος είναι ο μηχανισμός, πώς συμμετέχουν στον ε, μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, θα ήθελα να δώσω έμφαση στο γεγονός ότι σίγουρα ως φορέας, ως διεθνής οργανισμός, ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσουμε στο μέλλον το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Αυτό είναι σαφές, γιατί θα αντιμετωπίσουμε όλο και συχνότερα και όλο και περισσότερο αυτές τις παραλλαγές των ακραίων καιρικών φαινομένων. Ε, τέτοια φαινόμενα έχουν διαπιστωθεί σε όλες τις χώρες συμπεριλαμβανομένης και της δικής μου. Επομένως χρειαζόμαστε ένα πλάνο, ένα σχέδιο, μια στρατηγική για να ενισχύσουμε, να εφαρμόσουμε μηχανισμούς πολιτικής προστασίας και να τους προϊκοδοτήσουμε με περισσότερα χρήματα. Τώρα για την κυβερνοασφάλεια. Να σας πω ότι πρόσφατα συναντήθηκα με μιας οργάνωσης εδώ στις Βρυξέλλες η οποία ασχολείται και με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια, με τις ασφάλειες ε, και με την ασφάλεια γενικότερα. Υπάρχουν δηλαδή εταιρείε που ασφαλίζουν για κυβερνοκινδύνους και ταπεινά προσκαλώ όλους εσάς ε, τη 10η του Οκτωβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου θα διοργανώσω ένα μεγάλο συνέδριο για το πώς καταπολεμείται ο, καταπολεμάται ο κυβερνοκίνδυνος και ο ρόλος της ασφάλειας για την καταπολέμηση ε, των ε, κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Ευχαριστώ πολύ χρήσιμο η κυρία Σόφκο παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν έχω πολλές ερωτήσεις. Ήθελα να σας συγχαρώ για το έργο σας. Στη Βοσνία Ρεζεγοβίνη, στη Σερβία το 2015 βοηθήσατε πάρα πολύ σε αυτό το τεράστιο πρόβλημα με τις πλημμύρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έδωσε την απάντηση που της αναλογούσε σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Και σε, αυτή την τρομερή κρίση φάνηκε πώς, ε, ε, πόσα πολλά μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη συντονισμένη της δράση, κάτι το οποίο δέχθηκαν πολύ καλά οι πολίτες όλων αυτών των χωρών. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο παράδειγμα. Το ερώτημα είναι τι μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε να συνεχίσετε την ε, καλή σας δουλειά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, αφού δεν ζητά κάποιος άλλος το λόγο, ε, να είναι αυτό το τελευταίο ερώτημα και να δώσω το λόγο στην κυρία Βαλεάν. Ναι, θέλω κι εγώ κάτι να πω. Συμφωνώ με σας κυρία Ζόφκο. Τα επιχειρησιακά κόστη δεν χρηματοδοτούνται και είναι πρόκληση. Αυτό λέτε εσείς. Όμως, τι χρειάζεται για να χρηματοδοτηθούν τα επιχειρησιακά κόστη. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό αφού εδώ είναι οι θύνοντες που λαμβάνουν τις αποφάσεις. Αυτό είναι μια ερώτηση που έχω εγώ να απευθύνω στον ομιλητή. Δεύτερον, θεωρείτε ότι το Brexit θα έχει αντίκτυπο στην εύρυθμη λειτουργία του κέντρου αντιμετώπισης έκτακτων ε, αναγκών. Και τρίτον, έχετε εμπλακεί Έχετε ασχοληθεί με το μεταναστευτικό, θα σκοπεύετε να ασχοληθείτε και αν ναι με ποιο τρόπο. Ευχαριστώ. Αυτές είναι οι τελευταίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Λούχνερ. Ευχαριστώ. Να σας πω καταρχάς ότι στην νομοθεσία προβλέπετε ότι μια υποψήφια χώρα είναι συμμετέχουσα χώρα του μηχανισμού. Αυτό κάνουμε για τους γειτονές μας. Έχουμε 28 κράτη-μέλη συν άλλα 6 κράτη που αποτελούν μέρος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Ή είναι χώρες προσχώρησης υποψήφιες που είναι στην προενταξιακή διαδικασία. Η Τουρκία λοιπόν είναι μέρος του μηχανισμού και εκτός και αν αποφασίσουμε θέματα που έχουν να κάνουν με την νομοθεσία ή τον προπολογισμό ή εκτός και αν ψηφίσουμε για το πρόγραμμα εργασιών, εκτός από όλα αυτά δηλαδή, για όλα τα υπόλοιπα, οι συμμετέχουσες γειτονικές χώρες έχουν θέση γύρω από το τραπέζι. Τώρα, ειδικά για την Νότιο Ευρώπη, Έχουμε χρηματοδότηση από το προενταξιακό ε, χρηματοδοτικό εργαλείο για τις πλημμύρες, για παράδειγμα, για χώρες της Βαλκανικής και προσπαθούμε να αναπτύξουμε μια ισχυρή διμερή σχέση, να οικοδομήσουμε δεξιότητες, ικανότητες εντός αυτών των χωρών. Είναι μια σχετικά αργή διαδικασία, υπερβολικά αργή ε, ε, κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι θέμα ανθρωπίνων πόρων. Για να γίνει κάτι καλά πρέπει να το κάνουν οι άνθρωποι και πρέπει να είναι καλός ο διάλογος με τους ανθρώπους. Φυσικά, Συμμετέχουν όλες αυτές οι χώρες στις ασκήσεις, ε, στα προγράμματα κατάρτισης, επιμόρφωσης, εκπαίδευσης. Ε, οι χώρες γειτονίας είναι οι χώρες που βρίσκονται γύρω από τη λεκάνη της Μεσογείου, τα Βαλκάνια αλλά και η Ουκρανία. Ενθαρρύνονται όλες αυτές οι χώρες να συμμετάσχουν. Και όταν ενεργοποιούμαστε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, πριν από 1,5 χρόνο η Αλβανία ενεργοποίησε το μηχανισμό για τις πλημμύρες. Προσπαθούμε όταν αποστέλουμε μία ομάδα πολιτικής προστασίας για να δράσει επιτόπου, να αξιοποιήσει την ευκαιρία για να οικοδομήσει επίσης ικανότητες και δεξιότητες επιτόπου. Δηλαδή ακόμα και όταν ανταποκρινόμαστε για να έχουμε πρόληψη ή ετοιμότητα, ε, ε, ενισχύουμε τις αρχές και συνοψίζουμε τις τοπικές αρχές τα βασικά σημεία της έκθεσης τα οποία μπορούν μετά στη συνέχεια να χρησιμοποιούν και μόνοι τους. Σε κάθε περίπτωση σας ευχαριστώ θερμά. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πεδίο. Παλιότερα εργαζόμουν στο τομέα της νομοθεσίας για τις χημικές ουσίες, όπου τα πράγματα ήταν πολύ πιο περίπλοκα και πολύ πιο δύσκολα. Ε, με δύο λόγια όμως θέλω να πω ότι είναι ένας τομέας πολύ σημαντικός, όπου θα έλεγα με πολύ μικρό κόστος έχουμε απτό αποτέλεσμα ορατό σε όλους. Και αυτό είναι κάτι που μας λένε όλα τα κράτη-μέλη. Έχουμε αυτή την ανταπόκριση από την πλευρά τους. Κάθε φορά που ε, ενεργοποιείται ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας και τα κράτη-μέλη και οι τρίτες χώρες αμέσως αναφωνούν. Ο Θεέ μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο ένα μάτσο γραφειοκρατών που λειτουργούν και κλεισμένο το θηρών στις Βρυξέλλες, αλλά έχει ε, κάτι να δώσει. Άρα λοιπόν η πολιτική προστασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ε, κάτι το ορατό, το απτό, με χειροπιαστά, πολύ θετικά αποτελέσματα. Είναι κάτι που λειτουργεί πολύ καλά, διότι Σύμφωνα με την νομοθεσία, ο ρόλος τη Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής δεν είναι ούτε καν να συντονίσει, αλλά να διευκολύνει τον συντονισμό. Και εμείς αντιμετωπίζουμε και ε, αρχές που έχουν τους δικούς τους περιορισμούς χώρες που έχουν πολύ κεντρική διοίκηση και που σε εθνικό κεντρικό επίπεδο αποφασίζονται τα πάντα. Έχουμε να κάνουμε χώρες όπου είναι ομοσπονδιακά κράτη, όπου από το Σύνταγμα οτιδήποτε, οτιδήποτε δεν έχει να κάνει με την εθνική άμυνα είναι αρμοδιότητα αποκλειστική του εκάστοτε κρατηδίου, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα, η Αυστρία και ε, είναι πολύ δύσκολη η έβρεση ενός κοινού ε, παρονομαστή και γίνεται και συζήτηση στα κράτη-μέλη για τα κόστη και λοιπά θέματα. Εμείς προσπαθούμε να βρούμε επικοδομητικές λύσεις που να είναι αποδεκτές από όλους, διότι σε αυτό το τομέα ο κόσμος λειτουργεί εθελοντικά. Κανείς δεν υποχρεούται να συνεισφέρει και κανείς δεν εξαναγκάζεται να συνεισφέρει. Άρα χρειάζεται να διατηρηθεί η καλή βούληση, η καλή θέληση. Μπορεί να είμαστε πιο βραδείς με τις ε, συζητήσεις μας ακριβώς γιατί δεν υπάρχει καταναγκασμός. Ε, όταν όμως φτάνουμε σε συνένεση και είμαστε δημιουργικοί, τότε τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά καλά. Και φάνηκε αυτό και το 2015 και σε άλλες περιπτώσεις και περιστάσεις. Σαφής διαχωρισμός εργασιών για ενεργοποιήσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κάτι πάνω στο οποίο όλα τα κράτη-μέλη συμφωνούν. Και όταν πλησιάζουμε κοντά στο να χαρακτηρίσουμε ένα περιστατικό ως έκτακτη ανθρωπιστική βοήθεια, τότε ε, η χρηματοδότηση μερικές φορές ε, ε, καθίστεται αναλόγως είτε πιο εύκολη είτε πιο δύσκολη αλλά νομοθετικά υπάρχουν κάποια κολλήματα εκεί και καλό θα είναι να τα άρουμε δηλαδή μπορεί να υπάρξει βελτίωση της νομοθεσίας εκεί Τώρα, ως προς το Brexit και ως προς την αξιολόγηση κινδύνου, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια πολύ προχωρημένη χώρα. Έχουν τρομακτική εμπειρία και τεχνογνωσία ε, για την ανάλυση ε, κινδύνου. Άρα το Brexit θα έχει επίπτωση σε αυτό. Τώρα, ως προς τον ενωσιακό μηχανισμό πολιτικής προστασίας, είναι ένας μηχανισμός που ενεργοποιήθηκε για το μεταναστευτικό και ενεργοποίηση για την Ελλάδα ήταν η μεγαλύτερη που είχαμε και το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισέφερε ε, σημαντικά, σημαντικότατα. Αυτό ήταν και η μεγαλύτερη μας επιχείρηση. Και τι συνέβη. ήταν λίγο παραπάνω από τις πρώτες βοήθειες, με δεδομένο τον αριθμό των ανθρώπων και το μέγεθος της πρόκλησης, δεν δώσαμε περισσότερα. Δώσαμε απλά τις πρώτες βοήθειες και πέρασε νομοθεσία για τον μηχανισμό, το εργαλείο επίγουσα στήριξης, αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών. Και αν δείτε πώς ενεργοποιήθηκε αυτό το εργαλείο, Μόλις ενεργοποιήθηκε αυτό το εργαλείο, οι δικές μας παραδόσεις αγαθών μειώθηκαν. Γιατί τελικά όταν έχουμε τέτοιου είδους κρίσεις είναι πιο λογικό να δίνουμε χρηματοδότηση στο κράτος μέλος από το να μεταφέρουμε εμπορεύματα με αεροπλάνα και πλοία από όλα τα μέρη της Ευρώπης στην Ελλάδα. Σας ευχαριστώ, η Πρόεδρος, και εγώ σας ευχαριστώ ε, που απαντήσατε όλες τις ερωτήσεις παραμένουν κάποια κενά όπως είναι η εκένωση με τα, η διακομιδή των ε, υπηκών ευρωπαϊκών χωρών. Η κυρία Βαλεάν έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ κι εγώ. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Περιμένουμε το Σεπτέμβρη. Χαιρόμαστε διότι εργάζεστε πάνω στις εταιρικές σχέσεις, στην πρόληψη, σε θέματα κατάρτισης, επιμόρφωσης, όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα για να υπάρξει ένα στέρεος μηχανισμό για το μέλλον. Επομένως, κατά τη δική μου αξιολόγηση, ε, όλα αυτά τα οποία μάθαμε σήμερα είναι ενθαρρυντικά και στοιχειοθετούν την ανάγκη να στηρίξουμε την εργασία σας, το έργο σας. Επομένως θεωρώ και πιστεύω ακραδάντως ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι σύμμαχός σας πανίσχυρος εταίρος σας για την προσπάθεια ενίσχυσης των μηχανισμών συνεργασίας. Σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε σήμερα και να ευχαριστήσω και την Πρόεδρο της Επιτροπής για την αποκοινού συνεδρίαση. Και εγώ σα ευχαριστώ, λέει η κυρία Μακαέβαν. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους από την ε, Επιτροπή ΕΜΒΗ να τους δώσουμε ένα-δύο λεπτά για να αποχωρήσουν για να συνεχίσουμε με τις εργασίες της δικής μας Επιτροπής.